Uh, Καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση της 28ης Απριλίου της Επιτροπής μας. Η συνάντησή μας, η συνεδρίασή μας σήμερα θα διαρκέσει ως τις 12.30 το μεσημέρι. Το πρώτο σημείο είναι έκθεση από την Europol για την ε, έκθεση TISAT την κατάσταση για την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τάσεις που διαγράφονται. Το θέμα θα μας το παρουσιάσει ο κύριος Wainwright, διευθυντής της ε, Ευρωπόλ. Θα σας δώσω το ρόλο κύριε Wainwright για να παρουσιάσει την έκθεση αυτή και βεβαίως μετά θα έχουμε συζήτηση. Παρακαλώ, ακούτε την ελληνική καμπίνα, ακούτε την ελληνική καμπίνα, είμαστε στη διάθεσή σας. Στην ε, καμπίνα αριθμός 7, ακούγεται καλά η ελληνική καμπίνα, σας παρακαλούμε. terrorism situation in the EU. Uh, you have uh, today been circulated with uh, the copies of our report for this year. Um,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 And what legal safeguards would you consider necessary? Thank you, Sarah. Ms. About effectiveness as, as much as, as the dangers of discrimination. Thank you, Sarah. Mr. Borghesio. Grazie Presidente, signor Direttore, mi unisco anch'io agli elogi per l'attività svolta da Europol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 In the meantime, the representative of the President of the Council arrived, Mr. Valentin Dueras Jimenez. I will give you the floor, and afterwards I will ask the shadows for intervention. Thank you. Mr. Gracias, señora presidenta. Eh, Bueno, permítanme eh, que comience eh, manifestando en nombre de la presidencia española del Consejo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 Ευχαριστώ. Let's reopen our meeting. Uh, This meeting is a joint committee meeting with the Committee of Subcommittee of Human Rights and Αρχίζει η συνεδρίαση, από συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Η κυρία Χαουτάλα ψηφίζει αυτή τη στιγμή σε μια άλλη επιτροπή. Η κυρία Ζολή δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει εκ μέρους των επιτροπών που προανέφερα. Αλλά θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευχαρίστησή μας και την τιμή που έχουμε, που έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών δια τους πρόσφυγες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Πατερμοστά την προηγούμενη εβδομάδα που επανεξελέγεται όταν η Γενική Συνέλευση ψήφισε την ανανέωση της θητείας σας για τα πέντε χρόνια. Αναμφίβολα αναγνωρίστηκε ο επικοδημητικός ρόλος σας και τα ηγετικά σας προσόντα και εμείς είμαστε ιδιαίτερα, ιδιαίτερα ευτυχείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σας καλωσορίζουμε εδώ πέρα. Παρακαλώ, ακούγεται καλά η ελληνική καμπίνα, ακούτε καλά την καμπίνα αριθμό 7, τα ελληνικά. Θέλετε να μας κάνετε ένα νεύμα, να ακούγονται καλά τα ελληνικά στην αίθουσα σας, παρακαλούμε στη θέσή σας. Ένα νεύμα σας παρακαλούμε, να ακούγεται καλά η ελληνική Ευχαριστούμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και θα θέλαμε να υποφεληθούμε από την παρουσία σας για να μας εξηγήσετε κάποια πράγματα το πόσο δύσκολο θέμα σας απασχολεί όσον αφορά την πρακτική οργάνωση των ε, εργασιών μας. Α, βλέπω ήρθε η κυρία Χαουτάλα, κάτι θα έλεγα, την περιμέναμε να έρθει. Εάν συμφωνείτε, θα μοιραστούμε την ε, Προεδρία, κυρία Χαουτάλα. Μετά την ε, παρέμβαση του κυρίου Γκουτέρες, θα σας δώσω την Προεδρία για να ηγηθείτε των συζητήσεων. Λοιπόν, κύριε Γκουτέρες, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μας κάνετε την παρουσίαση του θέματός σας. Δηλαδή, πώς βλέπετε τα πράγματα σε θέματα πολιτικής ασύλου. Και βεβαίω οι συνάδελφοι μετά θα κάνουν σχόλια και θα υποβάλουν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Γκουτέρες. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν έχω υπάρξει ποτέ Ευρωβουλευτής, όμως υπήρξα βουλευτής επί 25 χρόνια στη χώρα μου και συμμετείχα ενεργά στα ευρωπαϊκά θέματα και υποθέσει. Είναι λοιπόν μεγάλη μου χαρά που έρχομαι ξανά εδώ. Αισθάνομαι πολύ οικία. Στο κοινοβούλιο αυτό πάντοτε υπήρχε μια σοβαρή δέσμευση για τα ζητήματα ασύλου και την προστασία των ατόμων που χρήζουν διεθνού προστασία. Χαίρομαι λοιπόν που μιλάω σε γνώστε του θέματο. Εάν ξέρετε τώρα τι μεταναστευτικέ τάσει όπω ισχύουν παγκοσμίω, θα ξέρετε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για την Ευρώπη και αφού σχολιάσω την εικόνα της Ευρώπης θα περάσω και σε κάποια σχόλια για το μέλλον. Εάν δούμε τώρα σήμερα τι συμβαίνει με τον αριθμό μεταναστών και τους καταναγκαστικά εκτοπισμένους θα δούμε ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι αριθμοί είναι περίπου σταθεροί. 60 εκατομμύρια πρόσφυγε σήμερα, μαζί με του Παλαιστίνιου πρόσφυγε, 27 εκατομμύρια άνθρωποι εσωτερικώ εκτοπισμένοι εντό των συνόρων τη χώρα του, λόγω ε, συγκρούσεων και πολλού ε, άσυλο σε όλη τον κόσμο, αλλά ιδίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αριθμοί παραμένουν σταθεροί, λίγο πολύ. Η σταθερότητα αυτή βέβαια τη τελευταία διετία από τη μια δείχνει ότι παραμένουν σταθερέ κάποιε συγκρούσει και από την άλλη ότι είναι δύσκολο να εξευρεθούν λύσει. Έχουμε καταβάλει σοβαρέ προσπάθειε από το πρόσφατο παρελθόν για να δώσουμε μεγαλύτερε δυνατότητε υποδοχή. Υποδοχής από τρίτε χώρε ε, και προ ε, νέε χώρε προορισμού και είχαμε και σοβαρά κίνητρα προς αρκετές χώρες. Η Τανζανία δέχτηκε να δώσει την επικότητα σε 60.000 Μπουρουντιανούς. Σε 160.000 μάλλον Μπουρουντιανούς. Οι οποίοι κατοικούσαν στη χώρα και τώρα έγιναν επισήμως πολίτες της ε, Τανζανίας. Επίσης ο οικειοθελής ε, παναπατρισμός προς την χώρα προέλευσης όταν επιληθεί μια σύγκρουση. Πέρσι είχαμε δυστυχώς μία μείωση. Μισές σε σχέση με τις επιστροφές, οι επιστροφές του 2009 ως προς το 2008. Πέρσι είχαμε λιγότερες από 400.000 επιστροφές σε σχέση με ένα εκατομμύριο που είχαμε το 2008. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιες συγκρούσεις παραμένουν και κάποιες ε, καταστάσεις που θα έπρεπε να έχουν βγει από τις συνθήκες αυτές έχουν οδηγηθεί πάλι σε συνθήκες αστάθειας, όπως ε, στο Αφγανιστάν. Και όπου βλέπουμε ότι είπατε η αρμοστία του αναγκάστηκε να αναλάβει δράση. Τώρα για τις επιχειρήσεις τις οποίες συμμετέχουμε. Βλέπουμε δύο ομάδες, δύο κατηγορίες καταστάσεων. Τη μία όπου έχουμε κρίσεις και από τις οποίες προέρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγε στον κόσμο. Θα έλεγα ότι μιλάμε για ένα τόξο κρίσο από την Νοτιοανατολική Ασία και περνώντα την Ασία από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν προ το Ιράκ και την Μέση Ανατολή. Ε, ακόμη και αν δεν σκεφτούμε το θέμα των, Παλαιστινιακών, των Παλαιστινίων προσφύγων, διότι άλλη ομάδα ε, έχει αναλάβει την προστασία αυτών των ε, πληθυσμών, επίσης το Σουδάν και μετά φτάνοντας προς την Αφρική, το κέρας τη Αφρικής και την Ιεμένη. Οι καταστάσεις λοιπόν αυτές φαίνεται ότι είναι αλληλοσχετιζόμενες. Όλες έχουν να κάνουν με ζητήματα ασφάλειας. Υπάρχει και ανθρωπιστική διάσταση και αφορούν την ασφάλεια όλου του πλανήτη. Πολλοί θεωρούν ότι οι τρομοκρατικές απειλές διεθνώς συνδέονται με πολλές από αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις αναχώρα και σε ένα βαθμό βρίσκονται στο κέντρο των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ του δυτικού κόσμου, όπως τον αποκαλούμε, και του μουσουλμανικού. Μιλάμε για σύγκρουση πολιτισμών. Και βεβαίω η παρέμβαση τη διεθνού κοινότητα για την επίλυση αυτών των κρίσεων είναι καθοριστική σημασία. Υπάρχουν και άλλε κρίσει στον κόσμο, κάποιε από αυτέ σε δραματικέ συνθήκε, όπω η λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο στην Κεντρική Αφρική. Αλλά με μία ε, διαφορά. Εδώ μιλάμε για απομονωμένε περιπτώσει με περιφερειακή διάσταση. Με δραματικέ ενδεχομένω ανθρωπιστικέ συνθήκε που δεν αφορούν όμω άμεσα την διεθνή ασφάλεια. Ή τουλάχιστον δεν διασυνδέονται μεταξύ του. Γι' αυτό τίνουμε και να τι παραμελούμε βέβαια αυτέ τι περιπτώσει και γι' αυτό και είναι όλο και πιο δύσκολο η διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση. Και για την πολιτική λύση των κρίσεων και για την ανθρωπιστική απόκριση στι ιδιαίτερε ανάγκε των πληθυσμών. όπως στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Μια χώρα που φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη αγνοούν και την ύπαρξή τη. Αλλά όπου υπάρχουν ακόμη πολύ σοβαρά προβλήματα. Μιλάμε λοιπόν για ένα πλαίσιο σταθερότητα που πρέπει να εξασφαλιστεί για του ε, εκτοπισμένου, αλλά και για κρίσει ανεπίλητε. ή και για περιπτώσει κρίσεων που έχουν επιληθεί, φαίνεται να έχουν επιληθεί αλλά αναθερμαίνονται οι συγκρούσεις. Υπάρχει ανασφάλεια, στάθεια και άλλες επισφαλείς καταστάσεις. In this context. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου είναι καθοριστική σημασίας. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί η Ευρώπη ανέκαθεν ήταν μια ήπειρο ασύλου. Και η δική μα παρέμβαση ήταν σημαντική πάντοτε για τη διεθνή προστασία. Αλλά γιατί η Ευρώπη δίνει και το παράδειγμα. Πρόσφατα συζητούσα με τον Πρωθυπουργό μια χώρα τη Ζωτανολικής Ασίας σε σχέση με την επαναπροώθηση πολιτών που εκδιώχθηκαν στη χώρα της προέλευσής του. Και όταν συζητήσαμε την κατάσταση, μου είπε γιατί με κατηγορείτε εμένα. Και οι Ευρωπαίοι τα ίδια κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τι εικόνα δίνει η Ευρώπη ω παράδειγμα. Ο κόσμος στρέφεται προς την Ευρώπη για τα θέματα ασύλου. Ό,τι γίνεται στην Ευρώπη τίνει να επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, βασική μας μέρημνα και ισχυρότερη διάσταση της συνεργασίας μας με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Επιτροπή, λόγω χάρη είχαμε χθε και σήμερα πολλές συναντήσεις με μέλη της Επιτροπής και θετική συνεργασία βεβαίως για τα ζητήματα αυτά. Η βασική μας λοιπόν μέρημνα είναι το γεγονός ότι σε μια περιοχή όπου κυκλοφορούν ελεύθεροι πολίτε από τη μια χώρα στην άλλη, εφόσον είμαι Ευρωπαίο πολίτη, μπορώ να πάω στο Βερολίνο λόγω χάρη χωρί να δείχνω το διαβατήριό μου στου ελεγκτέ, ούτε να αλλάζω χαρτονομίσματα. Αλλά σε αυτή την περιοχή υπάρχουν πολύ διαφορετικά συστήματα ασύλου από τη μια χώρα στην άλλη. Ένα συγκεκριμένο, τον άσυλο, που έρχεται από μια από τι χώρε που ανέφερα, Σομαλία, Αφγανιστάν ή την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, μπορεί να έρθει σε μια ευρωπαϊκή χώρα να ζητήσει άσυλο και κατά 98% μπορεί να απορριφθεί η αίτησή του σε μία χώρα, αλλά να πάει στη γειτονική και να έχει 70-80% πιθανότητες να αναγνωριστεί είτε ω πρόσφυγα είτε ω ε, άτομο που χρήζει άλλη μορφή ε, διεθνού προστασία. Στο πλαίσιο λοιπόν ενιαίου χώρου Έχουμε τόσα διαφορετικά συστήματα ασύλου και αυτό οδηγεί σε δυσλειτουργίε. Αποτελεί βασικό πρόβλημα για την προστασία των ανθρώπων και είναι και τεράστιο θέμα για την Ένωση. Διότι υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και είναι δύσκολο να ελέγξουμε τις ροές των ετούντων άσυλο και των προσφύγων, προσφύγων σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, οι πέντε προτάσεις τροποποίησεων οδηγιών που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δουβλίνο 2, Eurodac, συνθήκες υποδοχής, ε, απαιτήσει και διαδικασίες, πιστεύουμε ότι αυτές οι τροποποιημένες οδηγίες τι οποίε χαιρετίζουμε, θα είναι ένα θετικό βήμα πρόοδου για να οικοδομήσουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Και αυτό που μα απασχολεί είναι ότι οι προτάσει αυτέ βέβαια με κάποια δυσκολία προχωρούν και πολλά κράτη-μέλη προβάλλουν αντιρρήσει. Ω προ την πρόθεση των προτάσεων αυτών. Υπάρχουν συγκεκριμένα επιμέρου ζητήματα βεβαίω αλλά πέρα από αυτές τις μικρές διαφωνίες για την συνεκτικότητα του συστήματος και για την, το μέλλον του συστήματος όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Επίσης υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία με τη Frontex εδώ και θεωρώ σημαντικό στις συζητήσεις μας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα με το Ευρωκοινοβούλιο να ακολουθούμε πάντα το ίδιο σημείο αφετηρίας. Τα κράτη έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να διαχειρίζονται τα σύνορά τους με τρόπο υπεύθυνο έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τη δική τους μεταναστευτική πολιτική. Και είναι διαφορετικό βεβαίω το θέμα των μεταναστεύσεων στην Ευρώπη. Δεν καλύπτεται από, το δικό μου, το, από τη δική μου την εντολή στα καθήκοντα που έχω αναλάβει. Όμω, ω προ τη διαχείριση συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών πολιτικών, τα κράτη θα πρέπει να εξακολουθούν να παρέχουν προστασία στα άτομα που χρήζουν διεθνού προστασία βάσει του διεθνού δικαίου. Όλα τα συστήματα διαχείριση θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αλλά θα πρέπει να δίνουν και προτεραιότητα στην προστασία. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό λόγω των μετακινήσεων και των τάσεων των μετακινήσεων του πληθυσμού παγκοσμίω και το πώ ε, προωθούνται οι μετακινήσει αυτέ και από διακινητέ Επίσης βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι συγκρούσεις δεν πάβουν. Ε, και πολλές φορές πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη μόνο με, ο μόνος τρόπος να περάσουν με τα παράνομα αυτά δίκτυα. Η παράνομη λοιπόν διακίνηση ανθρώπων είναι κάτι που σαφώς ε, καταδικάζουμε. Αλλά υπάρχουν ακόμη και χειρότερες μορφές εμπορία ανθρώπων, γυναίκες και παιδιά που ζουν σε συνθήκες ε, δουλείας πλέον. Είναι αντικείμενα πλήρου και αποτρόπε εκμετάλλευση. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να αναλάβει κάποια δράση εδώ. Υπάρχει έλλειψη επενδύσεων. Ενώ με τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλε μορφέ οργανωμένου εγκλήματο, και αυτά βεβαίω μα απασχολούν ιδιαίτερω, όμω πρέπει πάντοτε να μην ξεχνάμε αυτή τη βασική μα μέρημνα. Ότι θα πρέπει να καταδιώκουμε και του εγκληματίε, αλλά να προστατεύουμε και τα θύματα. Όλα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία των προσφύγων στο σημερινό κόσμο. Πρώτη μας λοιπόν μέρημνα και μέγιστο ενδιαφέρον μας είναι να οικοδομήσουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Βεβαίως η κοινή γνώμη σε πολλές χώρες συγχαίει τη μετανάστευση με το άσυλο λόγω των διάφορων ανησυχιών περί ασφάλειας. Σήμερα οι συζητήσεις των πολιτικών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τα παρουσιάζουν τα θέματα αυτά, έχουν και κάποιες ξενοφοβικές τάσεις. Υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσει σε διάφορες χώρες. Και βεβαίως αυτό απειλεί την αποτελεσματικότητα των οργάνων προστασία ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μα απασχολεί και εμά ιδιαίτερω βεβαίω. Λίγα λόγια για την ύπατη αρμοστία. Προσπαθούμε εντατικά σε ένα πλαίσιο με πολλαπλές προκλήσεις παγκοσμίω. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιωθούμε και να κάνουμε και περισσότερα. Απλώς ανησυχούμε ότι δεν φέρνουμε πλήρως εις πέρα τους στόχους μας, και όπως ε, ορίζονται οι υποχρεώσεις μας από τις δημόσιες σχέσεις που έχουμε αναλάβει. Για την εσωτερική μας διοργάνωση, ξέρετε ότι το 40% της οικονομικής μας στήριξης προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο δεύτερος θεωρητής μας, συνολικά. Μιλάμε για σημαντική συνεισφορά εδώ και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη αυτή η συνεισφορά. Ξέρετε ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχουν και άμεσε ευθύνε για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προπολογισμού προφανώ. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει και το ανάλογο υπόλογο. Μια από τι δικέ μα πρώτε ανησυχίε είναι να διασφαλίσουμε ότι η συνεισφορά μα απευθύνεται ακριβώ στου ανθρώπου που πρέπει να φροντίσουμε και λιγότερο να καλύπτει τι ανάγκε του οργανισμού μα. Έχουμε καταφέρει όχι μόνο να διευρύνουμε τι δραστηριότητέ μα για του πρόσφυγε, αλλά να λάβουμε και μεγαλύτερε δεσμεύσει για του εσωτερικού εκτοπισμένου. Λόγω τη διεύρυνση και του συστήματο του ΟΗΕ και τη ανθρωπιστική κοινότητα. Καταφέραμε να αυξήσουμε κατά 50% τις δραστηριότητέ μα παγκοσμίω. Από 1,2 δι δολάρια περάσαμε σε 1,8 δι δολάρια δραστηριοτήτων, όγκο δραστηριοτήτων σε 4 χρόνια. Και είχαμε και 30% μείωση του προσωπικού μα στην έδρα μα. Έχουμε λοιπόν περικόψει το κόστο 41% του συνολικού μας κόστος το 2006 έφτασε το 95% τώρα. Όλο και περισσότεροι λοιπόν πόροι απευθύνονται στους σκοπούς προστασίας. Οι δύο τομείς όπου δίνουμε περισσότερη έμφαση και με, κάνουμε μεγαλύτερες επενδύσεις είναι η αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και το να πετύχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα και προστασία. Ιδίω στο πλαίσιο των ε, κοινών μετακινήσεων πληθυσμών. Επίση, για του πρόσφυγε στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Όλο και λιγότεροι βρίσκονται σε καταβλισμού και όλο και περισσότεροι περνούν στα αστικά κέντρα. Ο όγκο των μετακινήσεων αυτών είναι σημαντικό, μια σημαντική πρόκληση. Όπω θα ξέρετε, στι φτωχογειτονιέ του Ναϊρόμπι, του Κάιρο, ε, ε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα επαρκέ σύστημα προστασία. Ενώ ένα καταβλισμό προσφύγων είναι διαφορετικό πράγμα για πολλού άλλου λόγου. Επίση, επιδιώκουμε να καλύψουμε κενά στα συστήματα προστασίας μας για τους εσωτερικούς εκτοπισμένους. Αυτή η ανησυχία σήμερα είναι πολύ σημαντική, διότι εάν είναι κανεί πρόσφυγα σε ξένη χώρα, βρίσκεται υπό το σύστημα προστασία τη χώρα αυτή βάσει του διεθνού δικαίου. Και υπάρχει ένα οργανισμό η επατερμοστία με μια συγκεκριμένη εντολή που φροντίζει ότι όλα πρέπει να γίνονται ώστε να διασφαλίζεται η προστασία αυτή. Όμω, αν βρίσκεσαι εντό των σύνορων τη χώρα σου και σε πρόσφυγα, βρίσκεσαι υπό την ε, προστασία τη κυβέρνησή σου ουσιαστικά. Υπό την εξουσία τη κυβέρνησή σου. Και αυτό είναι μέρο και του αρχικού προβλήματο. Τώρα για το μέλλον. Διαβλέπουμε τρει τάσει που μα απασχολούν ιδιαίτερω βάσει των σημερινών συνθήκων. πρώτη τάση είναι η συρρήκνωση του ανθρωπιστικού χώρου. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παράσχουμε προστασία σε διάφορα σημεία του κόσμου λόγω ανασφάλεια βεβαίω. Τρει συνεργάτε μα σκοτώθηκαν στο Πακιστάν μόλι πέρσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό σε έναν οργανισμό όπω τον δικό μα, όταν μέσα σε ένα εξάμεινο σκοτώνονται τρει συνεργάτε μα στην ίδια χώρα. Και αυτό αφορά κατά τον τρόπο και όλε τι ανθρωπιστικέ οργανώσει είναι η ασφάλεια λοιπόν ένα πρώτο παράγοντο, έπειτα η κυβερνητική δράση. Το είδαμε στον Ταρφούρ, το είδαμε σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι κυβερνήσει δυσκολεύουν την ανθρωπιστική πρόσβαση. Και έπειτα το τρίτο είναι η δυσκολία σε κάποιε από αυτέ τι περιπτώσει να διακρίνουμε την στατιωτική παρέμβαση τη διεθνού κοινότητα και την ανθρωπιστική διάσταση τη παρέμβαση αυτή. Για παράδειγμα, οι διαπραγματευτέ ε, τη ειρήνη η τήρηση των συνδικών ειρήνη. Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουν αυτό οι συγκεκριμένοι συνεργάτε μα. Αυτό που γνωρίζουμε στην ύπατη αρμοστία είναι ότι είναι πολύ πολύπλοκη η εντολή μα. Είναι πολύ δύσκολο να διασφαλίσουμε προστασία στου πολίτες, στο Κονγκόλογο χάρη, που έπρεπε να προστατευτούν οι πολίτε, αλλά και να καταπολεμηθεί ο στρατό που, που ήταν αντιμέτωπος με του αντάρτε. Και αυτό γιατί λόγω των εσωτερικών συνθήκων τη χώρα χρειάστηκε να υπάρξει και μια μορφή ισορροπή μεταξύ των δύο δυνάμεων για λόγου ασφάλεια τη χώρα αυτή. Ήταν δύσκολο επίση να διακρίνουμε ποιο μέρο του ΟΗΕ διασφάλιζε συνθήκε ειρήνη σε κάποια χωριά και ποιο αποστατική άποψη και ποιο διασφάλιζε την προστασία των πολιτών. Συρρυκνώνεται λοιπόν ο ανθρωπιστικό χώρο. Και επίση κάποιε φορέ και οι συνεργάτε των ανθρωπιστικών οργανώσεων γίνονται και στόχο όσο και αν προσπαθούν να μείνουν πιστοί στις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, που είναι καθοριστική σημασία για το έργο, για το έργο τους παγκοσμίως. Έπειτα, οι προτεραιότητε για του ε, ανθρωπιστικού στόχου ε, χάνουν μέρο του κύρου του παγκοσμίω. Πριν από 10 χρόνια ε, συμμετείχα στην κυβέρνηση, στη δράση τη κυβέρνηση τη χώρα μου για την επίλυση τη κρίση στο Ανατολικό Τιμόρ. Όμω, ε, με τι συνθήκε που επικρατούσαν πριν 10 χρόνια θα έδινα διαφορετική απάντηση για τι δυνατότητε επίλυση του προβλήματο στη χώρα αυτή. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Βλέπουμε πάντω ότι η σειρά προτεραιοτήτων των ανθρωπιστικών οργανώσεων χάνουν πλέον ε, ένα μέρο τη σημασία του και κάτι που θα είναι σημαντικό και για τα μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι δύσκολο να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα της ανθρωπιστικής δράσης και να έχουμε και την απαραίτητη αναπτυξιακή στήριξη εδώ. Στον τομέα αυτό δεν νομίζω ότι επιτελούμε επαρκή πρόοδο. Διότι δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση από την πλευρά των ίδιων των χωρών, αλλά και υπάρχουν δυσλειτουργίε στον τρόπο που η διεθνή κοινότητα διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα. Και ένα τελικό σχόλιο για το μέλλον. Είμαστε μάρτυρες σήμερα νέων τάσεων για τους καταναγκαστικούς εκτοπισμού. Βεβαίως υπάρχει ανάλογη σύμβαση που ισχύει για τα θύματα των εσωτερικών συγκρούσεων, όμως η σύμβαση του 51, όμως υπάρχουν όλο και περισσότερε μετακινήσει παγκοσμίω λόγω των οικονομικών συνθήκων αλλά και άλλων λόγων. Εάν δείτε τις σημερινές τάσεις, την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, 9 δισεκατομμύρια το 2050, την ε, εξάπλωση των αστικών κέντρων. Το μεγαλύτερο μέρο του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει ω το 2050 σε αστικά κέντρα. Τι κλιματικέ αλλαγέ. Όλοι αυτοί οι παράγοντε δημιουργούν συνθήκε ανασφάλεια και οδηγούν σε μετακινήσει. Η έλλειψη νερού, η λειψιδρία δηλαδή, μετακινήσει των ανθρώπων. Όλα αυτά είναι προ... θέματα που αλληλοσυσχετίζονται και υπάρχει και συρρήκνωση ταυτόχρονα. Δυσκολίες για την ανάπτυξη. Όλα αυτά όχι μόνο γίνονται αλληλοσυσχετιζόμενα, αλλά συνδέονται και με την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα και γίνονται ε, αιτίε για την εκτοπισμό. δεν είναι σαφέ αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για τα ζητήματα αυτά. Κάνουμε κάποια πράγματα για τον επισητισμό, κάποια πράγματα για το νερό, κάποια πράγματα για του πρόσφυγε, αλλά ξεχωριστά. Δεν υπάρχει μια συνολική προσέγγιση για όλα τα προβλήματα από κοινού. Διότι, όπω είπα, είναι ελληνοσχετιζόμενα και γίνονται αίτια, τα βασικά αίτια για τον ιστορικό εκτοπισμό. Δεν μπορούμε να πειράξουμε τη σύμβαση του 51, γιατί πιστεύω ότι αν αποπειραθούμε κάτι θα γίνει χειρότερη από ό,τι ήταν τότε. Το ίδιο θα γίνει και με την ε, χάρτα των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Εάν τους ε, είχαμε αποπειραθεί να την απαναδιτυπώσουμε, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ θα διασφαλίσουμε την ε, προστασία του χρόνου. Θα γιορτάσουμε την 60η επέτειο της σύμβασης ε, του 51 και θα δώσουμε έμφαση στο θέμα των απατρίδων. Οπότε σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις ε, δράσεις και τη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ελπίζουμε το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξουν καθοριστικό ρόλο για να δοθεί μια σαφής απόκριση στα ζητήματα αυτά των ε, δύο εκτοπισμών, των εσωτερικών εκτοπισμών και να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες προστασίας παγκοσμίως σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκουτιέρες. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα, σημαντικά αλλά και θλιβερά τόσα μας είπατε. Αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι και λόγοι να εγκύψουμε στις τάσεις αυτές. Θα παραδώσω την διεύθυνση της συζητήσεως τώρα στην κυρία Χαουτάλα. Έχουμε πλήρωνε αγορητέ εγγεγραμμένου. Σας ευχαριστώ, λέει κυρία Χαουταλά. Εξ ονόματο της ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σα καλωσορίζω. Ευχαριστώ και την Επιτροπή ε, Θεμελιωδών Ελευθεριών που ε, διοργάνωσε την κοινή αυτή συνεδρίαση. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό των διασυνδεδεμένων φυσικών ορίων που αναπτύξατε και εσείς στην εξαιρετική ομιλία σας σας βεβαιώνω ότι στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εργαζόμαστε και για τις εξωτερικές σχέσει μας ενδιαφέρει όλο και περισσότερο αυτή η διασύνδεση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών της ε, μετανάστευση, της μετακίνησης πληθυσμών κλπ. Και είμαι βεβαία ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και για ε, θέματα εμπορίου ανθρώπινων όντων. Δεν θα παρατείνω ωστόσο ε, το χρόνο της συνεδριάσεως προσθέτοντας δικά μου σχόλια στα όσα είπατε. Θα καλέσω τα παρόντα μέλη να λάβουν το λόγο και έχω πρώτα την κυρία Αλφάνο. Ε, νομίζω ότι πρέπει να τεθεί όριο στον χρόνο αγορεύσεως. Ας πούμε δύο λεπτά, δύο λεπτά ως σύσταση. Ευχαριστώ. Και εγώ καλωσορίζω τον εκπρόσωπο της ΕΠΑ της Αρμοστίας Μας ικανοποιεί ιδιαίτερη παρουσία σας εδώ και ίσως να μας δώσετε και κάποιες απαντήσεις που να καθησυχάζουν. Τώρα, κάποιες ερωτήσεις εδώ στην Επιτροπή μας, εδώ στο Κοινοβούλιο, ήδη από το Σεπτέμβριο ενδιαφερθήκαμε για την πληγή που όλοι γνωρίζουμε των επανατρισμών. Ξέρουμε τι έγινε στις 29 και 30 Αυγούστου στην Ιταλία όταν 55 πρόσφυγες επαναπατρίστηκαν 75 πρόσφυγες ε, επαναπατρίστηκαν από την Ιταλία προς τη χώρα τους και ξέραμε ότι η πρόθεσή τους ήταν να ζητήσουν άσυλο στη χώρα μας. Ξέρετε ότι στις Σιρακούσες υπευλήθη μήνυση κατά του υπεύθυνου των συνόρων Ρονκόνη και του υπεύθυνου της ε, εθνικής ε, της δίωξης οικονομικού εγκλήματος ε, στον Δήμο αυτό που οδήγησε βεβαίως στην επαναπατρισμό των προσφύγων αυτών στη Λιβύη. Η Ιταλία τώρα επιδίωξε την επίτευξη διμερού συμφωνίας με τη Λιβύη και να θυμίσω εδώ ότι η Λεβή δεν έχει συνυπογράψει ποτέ τη σύμβαση της Γενέβη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει εδώ μια συμφωνία πλαίσιο και να την επιδιώξουμε ενεργά. Το ίδιο συμβαίνει και με το Πακιστάν στις διαπραγματεύσει, Μα ούτε το Πακιστάν έχει επικυρώσει την σύμβαση της Γενέβης. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία καθοριστικά για την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνίες και εφόσον είναι εδώ παρόν και το Συμβούλιο, αυτό που θέλω οπωσδήποτε να ρωτήσω είναι Γιατί δεν ενημερωθήκαμε για τις συζητήσει που γινόντουσαν μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τότε προέδρευε η Σουηδία και των ε, επιευθύνων του Πακιστάν και της Λιβύης. Τους ε, τελευταίους μήνες Ο εκπρόσωπος στην Ιταλία κατήγγειλε όχι μόνο αυτό που συμβαίνει στις φυλακές της Λιβύης όπου φτάνουν αυτοί οι άτυχοι άνθρωποι που πολλές φορές προσπαθούν να ξεφύγουν από θρησκευτικού διωγμούς, από διωγμούς κατά των πολιτών στις χώρες τους και από διδακτοτερικά καθεστώτα. Εκεί καταλήγουν αυτοί οι επαναπατριζόμενοι και πολλές φορές ε, είμαι σίγουρο ότι καταφέρουν να μιλήσουν με υπαλλήλου του ΟΗΕ οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο επιβαρυντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να επιδιώξουμε αυτέ τι συμφωνίε πλαίσιο με χώρε που δεν έχουν ε, κυρώσει την Σύμβαση τη Γενέβη. και να γίνει κάποιο θετικό βήμα για υποθέσεις όπως αυτή που είναι πολύ σημαντικές. Μιλήσατε εδώ για συνθήκες δουλείας στις οποίες ζουν κάποιες φορές τα άτομα αυτά. Να το δούμε λοιπόν αυτό στο επίπεδο της Επιτροπής μας. Γιατί δεν έχουν προχωρήσει αρκετά αυτές οι συμφωνίες πλαίσιο. Γιατί βρισκόμαστε σε τέτοια βεβαιότητα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν γνωρίζουμε ούτε καν τι συζητιέται. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Αλφάνο. Ακολουθεί ο κύριος Κούριο. Ας ακούσουμε μετά από μια πρώτη σειρά τριών ερωτώντων τον ε, εκπρόσωπο του είπα του αρμοστή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, παρουσία του είπα του αρμοστή. Πρέπει να πω ότι εγώ ήμουν στην αντιπολίτευση όταν ήταν ε, Πρωθυπουργό ο Αντώνιο Γκουτέρε στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζω τις εξαιρεστικές του ικανότητες και τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του στον ΟΗΕ και θα ήθελα να χαιρετήσω τον συμπολίτη μου. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την ειλικρίνη με την οποία μας μίλησε, κυρίως για τα σχέδια για το μέλλον και για τον ειλικρινή τρόπο και για τις επικρίσεις που έκανε και για τη διεθνή κοινότητα και για την Ευρώπη. Σωστά η έκθεσή σας ε, υπογραμμίζει κάποιες αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως όλοι θέλουμε και να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Η Κομισιό ε, θέλει να ακολουθηθεί αυτή η κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν ε, μεγάλες αντιστάσεις από τα κράτη-μέλη. Εμείς με την ε, ψήφο μας εγκρίναμε την έκθεση του Ρούι Ταβάρε, του συμπατριώτη μας επίσης στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, για να προχωρήσει το θέμα των προσφύγων. Δεν είναι εδώ διότι πίνει στην και αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να σπάσουμε αυτή την αντίσταση των περισσότερων κρατών της Ευρώπης. Πρέπει να σας πω ότι ο διάλογος το Συμβούλιο δεν ήταν εύκολος και κυρίως με τους εθνικούς εκπροσώπους. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον κύριο Επίτροπο ότι η υποστήριξη της ΥΠΑ της είναι πολύτιμη. Όχι μόνο σε ειδικά θέματα, διότι στην έκθεση Βάρες λέγεται ότι η Ευρώπη έκανε πάρα πολύ λίγα πράγματα για θέματα επανεγκατάστασης προσφύγων και ε, ε, μας υπενθύμησε το 40% των ε, πόρων του που πηγαίνουν από την δική του ε, οργάνωση των Ηνωμένων Έθνη για τους Πρόεδρους στην Ευρώπη. Μας λέγει λοιπόν η έκθεση αυτή ότι κάνουμε πάρα πολύ λίγα πράγματα στην Ευρώπη παρά τις ευθύνες που έχουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να συνεχίσετε να ασκείτε πιέσεις και να μας βοηθήσετε τεχνικά. Και βεβαίως, εάν έχετε να μας πείτε ε, κάτι πιο συγκεκριμένο και να πιέσετε ακόμη περισσότερο στο Κοινοβούλιο, είναι δεχτό και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοέλιο, ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο Κάρλος. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκουτέρες για την παρέμβασή του και για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει για τους πρόσφυγες κάθε φορά είναι και πιο σαφές στην Επιτροπή μας ότι οι ετούντες άσυλο και διεθνή ε, προστασία είναι όλο και περισσότερο και πρέπει κάτι να κάνουμε για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Όλοι γνωρίζουμε το ε, πρόγραμμα της Χάγης όπου έχουμε εναρμοσμένες πολιτικές σε άλλα θέματα και θα ήθελα να έχουμε και μια ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να έχουμε και μια τέτοια πολιτική στην Ευρώπη χωρίς τη συνδρομή της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών. Εσείς μιλήσατε για τη συνεργασία με τη Frontex. Πέρσι εμείς πήγαμε στη Βαρσοβία και στη Βαρσοβία μας είπαν επίσης ότι υπάρχει συνεργασία με την ΥΠΑ Αρμοστία του ΟΗΕ αλλά θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα Πώς έχει η συνεργασία σας με τη Frontec. Δεύτερον, εμείς την προηγούμενη θητεία πρέπει να πω ότι επισκεφθήκαμε κάποια κέντρα κράτησης στην ε, Γαλλία, εκεί που κρατούνται κάποιοι μετανάστες, όπως λέμε στα ισπανικά οι και οι θήτες. Και σε κάποια από αυτά είναι παρούσα η υπατιαρμοστία, σε άλλα όχι. Πείτε μου συγκεκριμένα, ποια είναι η παρουσία σας και ποια είναι η ανεκτικότητα των αρχών των κρατών μαλών, μελών συγγνώμη, και σε κάποια τέτοια διοικητικά κέντρα κράτησης δεν επιτρέπεται, είναι απούσα η ύπατη αρμοστία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντίας Θα ήθελα τώρα να στραφώ στον υπατορμοστή και να προσθέσω το εξής. το νέο ερευνητικό πρόγραμμα για την ε, η οδηγία για το θέμα του ασύλου είναι για μας ένα πάρα πολύ σημαντικό βοήθημα. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να απαντήσετε σε αυτούς τους τρεις συναδέλφους καταρχάς. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν μιλώ Ιταλικά, θα σας απαντήσω στα Αγγλικά. Στην ε, αξιότιμη Ευρωβουλευτή κυρία Αλφάνο Αυτό που τονίσατε είναι πράγματι η βασική πτυχή για την προστασία στην Ευρώπη. Δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ιασδήποτε υποδιαπραγμάτευση συμφωνίας. Ωστόσο, εμείς μιλήσαμε καθαρά σε σχέση με τις πτυχές αυτές, με την έννοια ότι είπαμε ότι είναι σημαντικό η αδίποτε συμφωνία με τρίτο μέρος να σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο και κυρίως την Σύμβαση του 1951. Αυτά που είπατε είναι σωστά και σημαντικά, γιατί στην σημερινή κατάσταση και ιδίως σε σχέση με την Λιβύη δεν υπάρχουν εγγυήσεις προστασίας που χορηγείται σε ε, πρόσφυγες που εμπίπτουν στι κατηγορίε προσφύγων τη ε, συνθήκη του 1951. Δηλαδή, καμιά φορά το γεγονό ότι ο ύποτο αρμοστή είναι παρόν στη Λιβύη προβάλλεται ω λόγο για, να, για τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει λόγος να μην αποστέλλονται πίσω στη Λιβύη. Όμως εκεί η παρουσία μας δεν αναγνωρίζεται ε, εκ του νόμου, δεν υπογράφει την συνθήκη του 51 η Λιβύη και η πρόσβασή μας δεν είναι τακτική, για παράδειγμα, σε στρατόπεδα προσφύγων. Καμιά φορά γίνεται, καμιά φορά δεν γίνεται. Και δεν έχουμε και τη δυνατότητα πλήρους παρέμβαση. Καμιά φορά έχουμε τη δυνατότητα μέσω κάποια μη κρατική οργάνωσης με την οποία συνεργαζόμαστε να αποφύγουμε, για παράδειγμα, να αποσταλούν πίσω στην Ερυθρέα κάποιοι ε, από εκεί αλλά σε άλλε περιπτώσει δεν μπορούμε. Άρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επαναπατρισμού στη Λιβύη διότι μπορούν δίθεν να δοθούν εγγυήσει προστασία. Βέβαια η κατάσταση είναι διαφορετική σε άλλα πλαίσια με άλλε χώρε. Ωστόσο είναι σημαντικό να διευκρινιστούν αυτά. Σε οποιαδήποτε συμφωνία γίνει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λιβύη, γνωρίζω πόσο δύσκολε θα είναι οι διαπραγματεύσει αυτέ, είναι πολύ σημαντικό πάντω να ληφθούν υπόψη οι ενισχύσει αυτέ περί την προστασία. Ευχαριστώ τον κύριο Κοέλιο για τα ευγενικά του λόγια. Ε, έχουμε συνεργαστεί σε συνθήκες φιλίας ως τώρα. Τον ευχαριστώ λοιπόν για την παρέμβασή του και για τον κύριο Ντίας Δεμέρα. Νομίζω ότι και οι δύο παρεμβάσεις αναφέρονται σε ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει εθνική λύση για τα θέματα ασύλου. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατόν να ευρεθούν εθνικές λύσεις για τα προβλήματα ασύλου. Τα κράτη όμως συνεχίζουν να προσδίδουν μεγάλη σημασία στην εθνική κυριαρχία. Και έτσι έχουμε μία αμφισημία. Το κάθε κράτος θέλουν να κρατήσουν ως κρατικό, εθνικό θέμα, το θέμα ασύλου. Απ' την άλλη είναι σαφές ότι ένα τέτοιο πρόβλημα δεν θα εξεύρει λύση παρά μόνο εάν αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Έτσι, έχουμε άτομα τα οποία μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη ανάλογα με τα συστήματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε χώρα και ανάλογα με το που θα βρουν, αν είναι δυνατόν, ε, προστασία. Και βεβαίως στο δρόμο τους βρέσκουν και λαθρεμπόρους και ανθρώπους οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται και καμιά φορά μπερδεύονται και αυτοί οι οποίοι καλή την πίστη ζητούν άσυλο και αυτοί οι οποίοι θέλουν να υποφεληθούν είναι οι οικονομικοί πρόσφυγες ή κάτι το παρεμφερές. Και το μήνυμά μου είναι πολύ σαφές για τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι οι κύριοι ευρωβουλευτές παρεμβαίνουν και στην πολιτική των κρατών τους. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει συνεκτική στρατηγική και συνοχή σε ό,τι κάνουμε στην Ευρώπη. Να, από του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου που θα πρέπει να προβλεφθεί και θα πρέπει εδώ βεβαίω να προβλέψουμε και τη διάσταση τη διεθνού συνεργασία και για τη Frontex. Υπάρχει. Πάρα πολύ σημαντική συνεργασία για θέματα όπως σχεδιασμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, αλλά εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στις επιχειρήσεις της Frontex επιτόπου. Και μπορεί η Διευθύντρια, αν θέλει να προσθέσει κάτι, έχουμε πρόσβαση, όπως σας είπα, σε κάποια θέματα, αλλά όχι στις ε, τρόπο με τον οποίο ε, κάνει τις επιχειρήσεις ε, επιτόπου η Frontex. Και βεβαίως η παρέμβαση ανάλογα με την χώρα είναι διαφορετική. Τώρα, στα θέματα των κέντρων ε, πρέπει να πω ότι έχουμε πρόσβαση σε κάποιες από αυτές. Υπάρχει και παρουσία ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και βεβαίως εμάς μας ενδιαφέρει το οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Εμείς πιστεύουμε ότι για τους ε, ετούντες άσυλο η κράτηση θα πρέπει να είναι η εξαίρεση του κανόνα. Όταν όμως υπάρχει κράτηση θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το γεγονός ότι κάποιος είναι υποκράτηση δεν θα πρέπει να δυσχεραίνει την πρόσβαση στις διαδικασίες για να επιληθεί το κάθε πρόβλημα. Θα ακολουθήσουν η κυρία Λάτφορντ, Έρστα και Κέλλερ. Πρώτα η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ. Και καλωσορίζω τον υποταρμοστή. Συμφωνώ με τον Κάλλος Κουέιο και δεν είμαι βέβαια και στην εθνική σας αντιπολίτευση. Πέραν αυτού ωστόσο γνωρίζετε βεβαίως την εκτίμηση που έχει το Κοινοβούλιο για το αξίωμα του είπα το αρμοστή. Θα ήθελα πολύ να έχουμε τακτικές επαφές, να μας ενημερώνετε και να άλληλο ενημερωνόμαστε για διάφορες αλλαγές της νομοθεσίας και διόλου μην διστάζετε να αναμειγνύεστε στην νομοθετική μας διαδικασία. Είναι σημαντικός άλλωστε ο ρόλος προτύπου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευγενός αλλά με σταθερό τρόπο μιλήσατε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί επιδείνωση του πλαισίου μας υποδοχής και προστασίας ετουμένων άσυλο. Βέβαια, από την άλλη μεριά, αυτό δεν σημαίνει ότι καθένας που έρχεται και ζητάει άσυλο πρέπει και να αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, αλλά έχουμε χαμηλότερο όγκο ετουμένων ασύλο, άσυλο τώρα στην Ευρώπη από ό,τι είχαμε πριν από 10 χρόνια. Αυτό αποτελεί σοκ για μένα και δείχνει πόσο καταβαραθρωμένα στην πραγματικότητα τα συστήματά μας. Και αποτέλεσμα είναι τα διαφορετικά ποσοστά, οι διαφορετικές αναλογίες αναγνώρισης που αφήνουν χώρο σε λαθρεμπόρους, σε δουλεμπόρους και ούτω καθεξής. Εν τέλει δηλαδή φτάνουμε να έχουμε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Όλοι τελικά χάνουμε διότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, διότι μεμφόμαστε τους ε, πρόσφυγες ως ε, ότι δήθεν έρχονται για να εποφεληθούν από την κοινωνική προστασία, από τις κοινωνικές ασφαλίσεις μας και ούτω Εγώ συμφωνώ πάντως μαζί σας ότι πρέπει να συνεργαστούμε ώστε του χρόνου που είναι 60η επέτειο της συνθήκη του 1951 και όπου τέλος πάντων 6 δεκαετίε μετά ίσως να χρειάζεται κάποιον εξυγχρονισμό αλλά από την άλλη μεριά είναι επικίνδυνο, συμφωνώ μαζί σας, να ανοίξουμε τον... την πηξίδα αυτής τη Πανδώρα, διότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε μέρη και ήδη η Βρετανική κυβέρνηση μιλούσε για ανανέωση της συνθήκης προδεκαετίας και δεν μου άρεσε. Ίσως χρειάζεται να συγκριθεί ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, με τις αιτίε δηλαδή που οδηγούν στον βιοεκτοπισμό, με τον ίδιο τρόπο όπως ασχολήθηκε και με την κλιματική αλλαγή, που είναι και ένας από τους λόγους βέβαια έμεσα που προκαλεί βιοεκτοπισμό. Μπορούμε να μιλήσουν και για την μετανάστευση που συνδέεται βέβαια και με την ε, νόμιμη μετανάστευση ή με την έλλειψη διάβλων για νόμιμη μετανάστευση, καναλιών δηλαδή όπου που να περνάει η νόμιμη μετανάστευση. Πέστε μας λοιπόν ειλικρινά, εάν η Ευρώπη κάνει ή δεν κάνει τα σωστά πράγματα. Και εγώ σέβομαι όπως, θα σέβομαι, σεβόμουν και πάντοτε τις συμβουλές σας, και επίσης το εάν έχει πρόσβαση ε, ο UNHCR στις επιχειρήσεις της Frontex, αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Δεν έχουμε πρόσβαση στη Λιβύη ή και δεν έχετε εσείς πρόσβαση στη Λιβύη. Δεν έχετε και πρόσβαση στις επιχειρήσεις της Frontex. Είναι εκπληκτικά τα πράγματα αυτά. Ξέρω ότι έχετε και επαφή με την Επίτροπο Μάλμστρομ που είναι και συνάδελφός μου και χρειάζεται να πείσουμε τις χώρες μέλη ότι δεν πρόκειται εδώ για καμιά γενεοδορία ή καλοκαρδοσύνη, αλλά είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα, να υπάρχει ένα σύστημα που να λειτουργεί καλά χορήγηση ασύλου. Και που εν τέλει θα μας βοηθήσει κιόλας και εμείς να ωφεληθούμε από τα προσόντα, τις δεξιοτεχνίες που φέρουν μαζί τους οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ και ζητούν άσυλο και μετά ενδέχεται να εγκατασταθούν και να δουλέψουν εδώ. Η κυρία Χαουτάλα. Σας ευχαριστώ κυρία Λάντφορντ. Χαίρομαι πολύ για την πρότασή σας για τον εορτασμό της 60ης επαιτίου. Είναι σωστό κύριε ε, είπατε αρμοστά να γίνει αυτό και με την ευκαιρία που είπατε. Η κυρία Έρστ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα Συγχαρητήρια στον κύριο Κουτιέρες για την επανεκλογή του που είναι πολύ σημαντική και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δυσχερές και επίπονο έργο σας. Θεωρώ πραγματικά απαράδεκτο να είναι τόσο περιορισμένες οι αρμοδιότητες του είπα του εκπροσώπου ώστε να μην του επιτρέπεται να είναι παρόν σε επιχειρήσεις Frontex. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο έχοντας συμφωνήσει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Frontex να υποχρεούται να τηρεί και τις αρχές προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θυμηθείτε την απόφαση που λάβαμε στην Ολομέλεια. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να ασκηθεί πίεση. Πρώτο σχόλιο αυτό. Δεύτερο τώρα. Λέχθηκαν πολλά και συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να υπάρξει και να ισχύσει κοινό δίκαιο ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μεμονωμένες εθνικές λύσεις. Αυτό είναι σημαντικό και σωστό. Και το λέμε καθημερινά. Η δική μου ανησυχία στην προκείμενη αυτή περίπτωση είναι ότι στην σχέση μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας, ασφάλειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενδέχεται να υπάρξει μια μετατόπιση υπέρ, θα έλεγα, της ασφάλειας ή ας πούμε της δίθεν ασφάλειας, θα έλεγα εγώ. Ανησυχώ δηλαδή ότι οι πτυχές της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων κινδυνεύουν να καταστούν δευτερεύουσα σημασίας κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να το ε, κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσουμε την πτυχή αυτή της ανάγκης προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μια τρίτη σκέψη που με καθοδηγεί είναι αυτές οι παναπροωθήσεις από την Ευρώπη ε, προς τρίτες χώρες και οι σχετικές συμφωνίες. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό, για παράδειγμα, να επαναπροωθούνται άνθρωποι που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, για παράδειγμα Κόσοβο, ε, για παράδειγμα η Ρώμα, που επανέρχονται, επαναπροωθούνται σε τέτοιες περιοχές σε τρομερά δύσκολες καταστάσεις. Ακόμα το Πακιστάν, το οποίο δεν έχει κυρώσει την συνθήκη της Γενέβης και όμως βγαίνουμε και συζητούμε τώρα και διαπραγματευόμαστε συμφωνία επαναπροώθησης με το Πακιστάν. Πράγματα δηλαδή ε, όπου θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, καθώς επίσης και τις συμβουλές που μπορείτε να μας δώσετε, γιατί ε, συζητούμε τώρα τις διαπραγματεύσεις αυτές ειδικά με το Πακιστάν και εμένα όπως είπα και πριν με ανησυχούν ιδιαίτερα. ευχαριστώ. Η Κέλλερ. Ευχαριστώ και για την παρουσία σας, τις ιδέες που ε, μας αναπτύξατε ερωτήσεις για τις νέες προκλήσεις που είπατε ότι θα αντιμετωπίσουμε. Ανθρώπων, για παράδειγμα, που καθίσταται πρόσφυγες λόγω αλλαγών του κλίματος. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ήδη. Τι νομίζετε όμως ότι πρέπει να γίνει σχετικά. Η αντιδράση που έχουμε μέχρι τώρα στην Ευρώπη, η ανταπόκριση δηλαδή, είναι επαρκής τι είδου προστασία νομίζετε θα πρέπει να χορηγήσουμε στα πρόσωπα αυτά που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν λόγω των συνεπειών των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε μπορέσει να ερευνήσετε καταγγελίες κατά της Frontex από το περσινό καλοκαίρι. Εμείς θέλαμε να ρωτήσουμε τον επικεφαλής της Frontex τι έχει κάνει σχετικά. Δεν απάντησε τίποτα. Εμείς θα θέλαμε να ελέγχουμε τι γίνεται. Διαρωτώ με αν έχετε κάνει έρευνες και αν μάθατε τίποτα. Για αν έχετε με κάποιο τρόπο άλλο μπορέσει να επηρεάσετε την κατάσταση εκεί. Είπατε ακόμη ότι προχωρείτε σε αναθεωρήσεις. Αυτό μου φαίνεται σημαντικό, αλλά ίσως είναι ένα βήμα, αλλά δεν είναι και επαρκές. Δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει στον δρόμο αυτό. Ρωτώ λοιπόν και εγώ, τι νομίζετε ότι ποια μορφή πρέπει να λάβουν αυτές οι αναθεωρήσεις οδηγιών. Ευχαριστώ. Ο ύπατος αρμοστής. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ την κυρία Λάντφορντ για τα σχόλιά της. Συμφωνώ άλλωστε με όλα τα σχόλια αυτά. Με τα σχόλια ε, στα οποία θέλω να κάνω μια υποσημείωση. Δεν έχουμε εντολή σε σχέση με την πολιτική μετανάστευση και βεβαίω οι χώρες μέλη έχουν ε, οι χώρες τέλο πάντων έχουν το δικαίωμα να ε, σχεδιάζουν και να ασκούν πολιτική μετανάστευσης. Ωστόσο υπάρχει μια πρόκληση ασυμμετρική, δηλαδή διακινούνται ελεύθερα τα κεφάλαια, διακινούνται ελεύθερα τα εμπορεύματα, όμως όχι τα πρόσωπα. Ε, ε, ακόμα και αν υπάρχει όλο και περισσότερο μια παγκόσμια αγορά εργασία. Όπως υπενθύμησε ο πρώην συναδελφός μου Κάρλος Κουέλιο, σοσιαλιστής, Εγώ ε, αναγκάστηκα και εγώ να μάθω ότι οι αγορές λειτουργούν και ότι κάποια στιγμή προσφορά και ζήτηση συναντώνται νομίμως ή δυνατόν παρανόμως εάν αυτό είναι απαραίτητο. Επομένως αυτά είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου θα αντιμετωπιστεί καλύτερα και η προστασία του πρόσφυγα. η χώρα μου πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία ε, γονιμότητας γύρω στο 1,4. Ο πατέρας μου πέθανε πέρσι στα 95 του και είχαμε βεβαίως και ανθρώπους στο σπίτι να τον φροντίζουν καθώς και τη μητέρα μου. Από τα 7 πρόσωπα που ασχολούνταν μόνο δύο ήταν Πορτογάλοι ή Πορτογαλίδες. Τα υπόλοιπα ήταν μετανάστες. Η μετανάστευση λοιπόν είναι σημαντική υπόθεση και για το ευρωπαϊκό μέλλον και είναι καλύτερα να τα ρυθμίσουμε εμείς παρά να τα αφήσουμε να τα ρυθμίζουν οι δουλέμποροι. Τώρα, για την κυρία Έρνστ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είχα χθε την ευκαιρία να συναντηθώ με την Επίτροπο Μάλμστρομ και διεξήγαγα ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ιδίως για την Frontex. Νομίζω ότι η εντολή της Frontex βρίσκεται υπό αναθεώρηση, υπό επανεξέταση τουλάχιστον. Ελπίζω ότι η εξέλιξη αυτή θα αποδειχθεί θετική. Σε ό,τι αφορά την ε, σχέση ασφάλειας και ελευθερίας. Νομίζω δεν υπάρχει αντίφαση. Εδώ νομίζω υπάρχει σύγκληση σε σχέση με το άσυλο. Δηλαδή, αν γίνονται, όταν θα γίνονται σωστά οι διαδικασίες του ασύλου, όταν δηλαδή οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται θα έχουν δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στις διαδικασίες αυτές, αυτό θα στηρίξει το κράτος. Από τις πιο, πιο δραματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε σε διάφορες χώρες του κόσμου είναι ότι τα νομικά συστήματα δεν είναι αρκετά φιλικά. Και ε, ε, επομένως αυτό τρέφει την παρανομία. Αυτό είναι αρνητικό όμως και για το κράτος. Πρόσφατα ε, μίλησα με την κυβέρνηση της Κένιας για τα σύνορα προς την ε, Σομαλία που υποτίθεται θεωρητικά ότι είναι κλειστά αλλά περνάνε χιλιάδες άνθρωποι πέντε χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν πρόσφατα χωρίς απολύτως κανένα screening είναι καλό αυτό για την ασφάλεια της Κένιας προφανώς όχι αν τα πράγματα γίνονταν με τρόπο ξεκάθαρο να περνούν δηλαδή νόμιμα τα πρόσωπα αυτά τα σύνορα ε, να ε, ελέγχονται αυτό θα μείωνε και τη δραστηριότητα των ε, ε, παράνομων διακινητών και ούτω καθεξής. Ε, όταν ένας τρομοκράτης δεν πάει να ζητήσει άσυλο, με άλλο τρόπο μπαίνει σε μια χώρα, διότι να πάει να ζητήσει άσυλο είναι περίπλοκη διαδικασία, όπως θα έχετε αντιληφθεί τώρα. Ακόμα και αν πάντως είναι περίπλοκο, περίπλοκη ιστορία. Η θέση μας σε σχέση με τον επαναπατρισμό το πρόβλημα τίθεται ε, στις απορρίψεις περιπτώσεων επαναβατισμού με τις απορρίψεις εκείνων των υποθέσεων που οδηγούν σε κάποιες φαιές ζώνες και εκεί και συζητούμε έχουμε κάποιες guidelines ε, σχετικά με χώρες προέλευσης που δεν γίνονται και πάντοτε σεβαστές μιλήσατε για το πρόβλημα των Ρώμα αυτό όμως υπερβαίνει ε, τις διαστάσεις του ασύλου πρόκειται για πολύ σοβαρές Υποθέσει ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ε, φανταστείτε, ήμουν προ λίγων εβδομάδων στον Καναδά. Ο μεγαλύτερο αριθμό ετουμένων άσυλο στον Καναδά σήμερα είναι οι Ρώμα οι οποίοι προέρχονται από μια ευρωπαϊκή χώρα. Και δεν θα πω πια ετούμενοι άσυλο στον Καναδά. Ε, Προφανώ πολλοί πάνε εκεί λόγω του ότι εκεί δραστηριοποιούνται οι παράνομοι διακινητέ. Αλλά είναι πολύ δυσάρεστο για την Ευρώπη ότι ο μεγαλύτερο αριθμός των ετουμένων άσυλο στον Καναδά είναι πολίτες μιας ευρωπαϊκής χώρας. Και πρόσφατα ο Καναδάς επέβαλε βίζα, προξενικές θεωρήσεις ε, για τις μετακινήσεις ορισμένων πολιτών κάποιες άλλες ευρωπαϊκής χώρας. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα το οποίο πρέπει όντως να αντιμετωπιστεί και δει αποτελεσματικά. Ε, ευχαριστώ επίση την κυρία Κέλλερ για τα όσα είπε σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Νομίζω ότι η αλλαγή του κλίματος πρέπει να εξεταστεί ως καταλήτης, ως επιταχυντής, ως επιταχυντής άλλων πραγμάτων. Πάντοτε βέβαια έχουμε φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, πλημμύρες. Δεν μιλώ για σεισμούς βέβαια, ούτε για τα ηφαίστεια που δεν είναι αλλαγή του κλίματος, αλλά αλλά έχουμε κυκλώνε, έχουμε τέτοια πράγματα. Αυτά πάντοτε γινόντουσαν. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα γίνονται πιο συχνά μεγαλύτερη ένταση και έχουν βαρύτερε συνέπειες ε, στους ανθρώπους. Για παράδειγμα, ξηρασία στην Ανατολική Αφρική. Πάντοτε είχαμε ξηρασία στο Σαχέλ. Τώρα όμως επιταχύνεται. Να λοιπόν, εδώ μπαίνει η αλλαγή του κλίματο μαζί με την ανασφάλεια σχετικά με τις προμηθείς τροφίμων, μαζί με την λειψιδρία και το καθεξής. Και αναγκάζει πολλούς να μετακινηθούν, διότι δεν υπάρχει τρόπος να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο επιδεινώνεται διαρκώς. Όμως προκαλεί και συγκρούσεις μεταξύ αυτών και των ε, αγροτών. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα αυτά ολοκληρωμένα και να βρούμε ολοκληρωμένες απαντήσεις. Δεν αρκεί να πούμε ότι υπάρχουν κλιματικοί εντό εγωγικών πρόσφυγες. Πρέπει να έχουμε μια συνολική, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως πιστεύω, νομίζω ότι ο αριθμός μέσων που διαθέτουμε για την προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι σημαντικός, αλλά χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το οπλοστάσιο που διαθέτουμε και να δημιουργήσουμε μηχανισμού συντονισμού μεταξύ χωρών, μεταξύ διεθνών οργανισμών και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξασφαλίσουμε πραγματική αποτελεσματική προστασία υπέρ των θυμάτων των ε, κινήσεων αυτών. Δυστυχώ αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ούτε καν μια στρατηγική για να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Και πολύ θα θέλαμε να δούμε να σημειώνεται κάποια κίνηση Νομίζω η κατάσταση που αναφέρατε έχει σχέση με την Ελλάδα. Προδημήνου βρέθηκα στην Ελλάδα και οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει σαφής δέσμευση της ελληνικής κυβερνήσεως για να υιοθετήσει αποτελεσματικό σύστημα χορήγησης ασύλου. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό το μοσαϊκό που σας ε, περιέγραψα προηγουμένως, η Ελλάδα βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, διότι είναι μία από τις εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παντίων ειδών ανθρώπων και βεβαίω και όσων ετούνται άσυλο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε πραγματικό σύστημα χορήγηση ασύλου. Τώρα υπάρχει, όπω είπα, πραγματική ειλικρινή δέσμευση από πλευρά τη ελληνική κυβερνήσεω. Εγώ πάντω θα ζητήσω η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την Ελλάδα στην προσπάθεια αυτή. Η Frontex είναι σημαντική στην περίπτωση αυτή, αλλά έχει και σχέση με την ε, πρόληψη της ε, επαναπρόθεσης, έχει σχέση με ε, κέντρα υποδοχής, έχει σχέση με την υποδοχή, την πρώτη υποδοχή των ετουμένων άσυλων που τώρα γίνεται από την αστυνομία, να υπάρξει ένα πραγματικό σύστημα, να αντιμετωπιστεί ο όγκος που έχει συσσωρευτεί των αιτήσεων ασύλου. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όπως είπα, εμείς διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πραγματικά έντονη διάθεση από πλευρά τη ελληνικής κυβερνήσεως να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να επιδειχθεί σημαντική η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ώστε να διασφαλιστεί η επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος που ε, είναι όπως είπα ε, η πύλη αυτή εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και μέσω της Ελλάδα, Όπως είπα δεν έχουμε άμεση πρόσβαση στις επιχειρήσεις που γίνονται. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε αν γίνεται το ένα ή το άλλο πράγμα. Γνωρίζουμε όμως ότι στα σύνορα αυτά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην επαναπρόθεση, στην επανεισδοχή. Για τις οδηγίες τώρα, είναι μια στιγμή. Η θέση μας είναι σαφής. Ε, παρακολουθούμε προσεκτικά τις ε, τροποποίησεις που προτείνονται Ορισμένες θεωρούμε ότι δεν είναι ε, ορθές. Πάντως το πιο σημαντικό είναι να γίνει μια κίνηση προς τα εμπρός. Και πιστεύουμε ότι οι ευρωβουλευτές μπορούν να συνεργαστούν με τις χώρες μέλη για να δούμε αν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Ορισμένες φορές με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι χώρες που έχουν στέρεα ε, συστήματα ασύλου προβάλλουν εμπόδια σε αυτή την ενοποίηση. Ενώ αυτή η ενοποίηση θα είναι και εποφελία τους, διότι είναι πολύ προτιμότερο εν τέλει ε, να υπάρξει ένα ενοποιημένο σύστημα, η, δεμή, η έλλειψή του δηλαδή αποβαίνει σε βάρος τους, εφόσον όσοι θέλουν να ε, ε, ζητήσουν άσυλο θα αποφύγουν τις χώρες όπου δεν υπάρχει πραγματικά στέρεο σύστημα ασύλου και θα πάνε σε αυτές που υπάρχει. Ελπίζω λοιπόν ε, εν προκειμένου να μπορέσετε κι εσείς να συμβάλλετε στην επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστούμε. Τώρα πρέπει να είμαστε πολύ εύστηροι με το χρόνο ομιλία. Οκτώ ομιλητέ, δύο λεπτά ο καθένα. Για να έχει το χρόνο και ο εύγλωτο και τόσο επαείων και υπεύθυνο αρμοστής να μα απαντήσει για τα θέματα αυτά. Κυρία Σαρτζεντίνη και μετά η κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ βρίσκομαι. Κύριε Γκουτέρες, έχω δύο ερωτήματα. Είπατε ήδη ότι η σύμβαση του 51 δεν έχει πολλές πιθανότητες να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως, επιτρέπει μεγάλο περιθώριο για τις αιτήσει. Η χώρα μου η Λετωνία για την ώρα έχει μόνο 16 με πρόσφυγες με το επίσημο καθεστώς. Όχι 60.000 ή 16.000, 16 μόνον. Και πέρα από τις αιματηρέ συγκρούσει που μπορεί να συμβαίνουν σε άλλες γειτονικέ χώρε δεν δεχόμαστε πρόσφυγες εύκολα. Έπειτα υπάρχει και η σύμβαση του 61 για τον περιορισμό των απάτριδων στη χώρα μου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα το θέμα αυτό. Το 71% των ε, ανθρώπων αυτών δεν έχουν ακόμη λάβει κάποιο επίσημο καθεστώς. Και δεν αρκεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λέμε ότι το θέμα της επικοότητας ε, θα λυθεί σε εθνικό επίπεδο. Το μόνο που έχει γίνει στην ε, Λετωνία με τη σύμβαση του 61 είναι κάποιες παρεμβάσεις από τον ΟΗΕ, τη δική σας την είπατε αρμοστία και άλλα διεθνείς φορείς, αλλά τίποτε το συγκεκριμένο. Δεν θα ήταν καλό λοιπόν να αναλάβουμε κάποια δράση για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ευχαριστούμε με την άδειά σας. Να πω και να επισημάνω ότι η κυρία Αντζελίλη πρέπει να φύγει για να προλάβει μια πτήση. Οπότε να ακούσουμε εκείνη αυτή αμέσω, εάν δεν σας πειράζει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους αλλά ιδίω τον ύπατο αρμοστή για την ε, παρουσία του και την προθυμία του να συζητήσει μαζί μας και για τα λόγια που μας είπε σήμερα εν είδη εισαγωγής. Νομίζω όλοι συμφωνούμε με όσα είπατε. Δηλαδή ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη να υπάρξει κατανομή των ευθυμών, ευθυνών. Σωστά μιλήσατε για μια συνολική προσέγγιση τη χρειαζόμαστε αυτή τη συνολική προσέγγιση. Αλλά ακόμη περισσότερο χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Δηλαδή τα 27 κράτη-μέλη να έχουν ένα σύστημα κοινό και εναρμονισμένο. Και όπως ορθώς είπατε, δεν μπορούν να υπάρχουν εθνικές λύσεις. Μπορεί να υπάρχει μόνο λύση ευρωπαϊκή. Είπατε και κάτι άλλο πολύ σωστό, ότι τα κράτη-μέλη κάνουν μάλλον ε, επικαλούνται την αρχή της κυριαρχίας τους, αλλά κάποιες φορές προκειμένου να επεκφύγουν κάποιων ευθυνών τους. Να προσθέσω εδώ λοιπόν ότι ίσως κάποια κράτη-μέλη να μπορούν να το επιτρέψουν αυτού του εαυτού του, να μην αναλάβουν τι ευθύνε του, δηλαδή, ενώ υπάρχουν άλλε χώρε όπω η δική μου ή όσε βρίσκονται στο ναι, φυλακή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σύνορα, που αναγκάζονται να αναλάβουν και περισσότερες ευθύνε από όσε τους αναλογούν. Άρα το συγκεκριμένο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω είναι ένα παράδειγμα από τη χώρα μου είναι ότι πολλές φορές έχουμε επικριτικά σχόλια για τις δημαρίες μας συμφωνίες και πιο συγκεκριμένα με την Λιβύη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει κανείς κριτική. Όμως ε, τα προβλήματα πολλές φορές είναι πρακτικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και εσεί ο ίδιος είπατε, και θα κλείσω εδώ, είπατε ότι με τη Λιβύη είχαμε σοβαρά προβλήματα. Είχαμε προβλήματα με τη Frontex, δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε έλεγχο, δεν ε, επιτυχάνουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Φτάνω, φτάνω στο ερώτημα. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, προτάσεις και καταγγελίε. Ιδάλω, ασκούμε μεν κριτική, αλλά στην πράξη ε, εμεί αυτό που χρειαζόμαστε είναι λύσει πρακτικέ. Ευχαριστώ. Κυρία Στρέλα είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με πολλούς συναδέλφους να καλωσορίσω τον υπατορμαστή, να τον ευχαριστήσω την παρουσία του και για την σαφέστατη και πλήρη παρουσία του και να τον συγχαρώ που επανεξελέγει. Πιστεύω ότι μπορώ να ερμηνεύσω το γενικότερο αίσθημα των Πορτογάλων και να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για την εξαιρετική εργασία που επιτελείται με τόση αφοσίωση. Και πάλι συγχαρητήρια για την νέα σας θητεία. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των νέων προσφύγων εξαιτία των κλιματικών ε, αλλαγών που αναφέρατε και σήμερα και άλλες φορές γιατί οι εμπειρογνώμονες χτύπησαν το καμπανάκι του κινδύνου έναντι στις ε, φυσικές καταστροφές, στις καταστροφές προκαλεί ο άνθρωπος και λαμβάνοντα υπόψη ότι υπάρχουν ε, δευμεύσει εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώ απέτυχε η διάσκεψη τη Κοπενχάγη και δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με την ε, προβλεπόμενη διάσκεψη του Μεξικού και δεν αρκεί να μειώσουμε το επίπεδο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Τι σύσταση μας κάνετε για να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις προς τα ευρωπαϊκά όργανα να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, όπως είπαμε, είναι πολύ πολύπλοκη και έχει να κάνει και με τον διάσταση την ε, παγκόσμια όλων αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ κύριε την Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοντά στα σύνορά μας θα αρχίσει να υπάρχει μια ομάδα νέων προσφύγων τη στιγμή την οποία το Ισραήλ άλλαξε τους κανονισμούς διαβίωσης στη Δυτική Όχθη κανόνες οι στρατιωτικοί τους επέτρεψαν πιο εύκολα να μεταφέρουν άτομα από την δική όχθη στη λωρίδα της Γάζας και να δημιουργήσουν και πιο πολλούς πρόσφυγες. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να χρησιμεύσει και εμάς. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο ε, Γκουτέρες, πώς αντιδρά σε αυτό το θέμα η Ευρώπη, πώς μπορεί να βοηθήσει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργούν αυτοί οι νέοι κανόνες. Εσείς τι υποδείξεις θα μπορούσατε να μας κάνετε για να αποφεύγονται αυτές οι ε, νέες ομάδες προσφύγων που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Φλότ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον είπα το αρμοστή που είναι εδώ. Πάντα τίνουμε να κάνουμε επικρίσεις προς τις ε, πολιτικές των κυβερνήσεών μας ε, ε, που σας υποδίζουν να κάνει δουλειά σας, αλλά επικρίνετε τους, επικρίνετε τους, θα τους το πούμε εμείς. Βλέπω στα δικά σας τα έντυπα ότι με ενδιαφέρον διαπιστώνουμε ότι η πρώτη χώρα που παράγει, αν θέλετε, πρόσφυγες είναι το Αφγανιστάν και η πρώτη χώρα που τους υποδέχεται είναι το Πακιστάν. Χθες ε, λέγαμε στην συζήτηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει διαπραγματεύσεις συμφωνιών με το Πακιστάν και είπαμε ότι θα πρέπει να το αποδεχθούμε, αποδεχθούμε αυτή τη συμφωνία. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι τι κάνετε εσείς ως είπατε αρμοστία στο Πακιστάν. Ποια είναι η άποψή σας για την δυνατότητα ναι ή όχι ε, να επαναπροωθηθούν σε αυτή τη χώρα Αφγανοί. Δεύτερον, και τελειώνω, στο δικό σας τον κατάλογο υπάρχει μία χώρα που είναι η Τουρκία ως μία χώρα προέλευσης ε, προσφύγων. Και εμείς θέλουμε να τη βάλουμε ως χώρα, ως Γαλλία, σε μία από τις δέκα σίγουρες χώρες. Και μέσα σε αυτή τη λίστα τι έχουμε ως πρώτη χώρα, την Κάνα. Μήπως ε, αυτή η έννοια της ε, ασφαλούς, της σίγουρης τρίτης χώρας αποτελεί τροχοπέδι και είναι μειονέκτημα το να είναι κανείς από αυτή τη χώρα για να μπορέσει να τύχει θετικής ε, ε, μεταχείρισης ως πρόσφυγας. Ευχαριστώ κυρία Γκυγιόμ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την ε, παρουσία σας, για τις δράσεις σας. Μιλήσατε για τους, τον αριθμό των ατόπων που είναι εκτουσμένοι στην Ευρώπη και είπατε παρόλα αυτό ότι σε σχέση με τον κόσμο ολόκληρο. Η Ευρώπη είναι Ήπειρος που απορροφά ένα μικρό μέρος. Ενώ πολλές χώρες λέγουν ότι τους έχουν κατακλείσει οι ετούντες άσυλο και οι πρόσφυγες. Πολλές φορές ε, βλέπετε ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται πολλές φορές δίνει λάθος ε, ε, εντύπωση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Θα ήθελα να σας κάνω δύο πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Είπατε και διαπιστώνουμε και εμείς ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ του θεωρητικού συστήματος για το άσυλο που έχει κάποια χώρα και της πρακτικής. Και βεβαίως υπάρχει και μεγάλη διάσταση μεταξύ ε, του εθνικού συστήματος και του ευρωπαϊκού. Βεβαίως, Δεν μπορεί κανείς να ζητήσει και να απαιτήσει, χτυπώντα το χέρι στο τραπέζι, όλοι να υιοθετήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα. Πρέπει κάθε χώρα να είναι πεπισμένη για να το κάνει. Επίση, υπάρχουν με τι διάφορε οδηγίε που συζητούμε αυτή τη στιγμή, όπω ξέρετε, διάφορα προβλήματα τα οποία θέλουμε να χειριστούμε οριζόντια. Όσον αφορά την ε, νομική συνδρομή, την προσωπική συνέντευξη που θέλουμε με κάθε ετούντα άσυλο αλλά δεδομένου ότι είναι αργά και δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, μπορείτε να μας μιλήσετε για τις δυσκολίες που έχετε βάσει συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Επίσης, να επανέλθω σε ένα άλλο θέμα, του κόστους. Ορισμένα κράτη-μέλη τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα του κόστους και πιστεύουν ότι για να ενεργήσουν γρήγορα εξαιτία του κόστους λένε, και αυτό είναι καρικατούρα, ε, πολλοί πρόσφυγες, ε, βιαστικά βρίσκουμε λίγοι, λίγοι πρόσφυγες, τα ε, προβλήματά τους θα λύνουμε με καλύτερο τρόπο. Το θέμα λοιπόν το οικονομικό, το ποιος αναλαμβάνει οικονομικά το βάρος της δαπάνης για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, πώς το βλέπετε, έχετε να πείτε. Ευχαριστώ ο κύριος Ρωσέτη, ε, Ευχαριστούμε τον είπα το αρμοστή για την προσέλευσή του σήμερα. Μπορούμε έτσι να έχουμε μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες δικές μου παρατηρήσεις. Και σε σχέση με κάποιες πολιτικές που αναπτύσσονται, στην Ευρώπη και όχι μόνο νομίζω. Κατά των δικαιωμάτων ασύλου ίσως. Θα ήθελα να θέσω και κάποια ερωτήματα. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα ασύλου γνωρίζουν μια υπαναχώρηση όπως και τα ζητήματα τα μεταναστευτικά. Φαίνεται να υπάρχει οπισθοδρόμηση και η στάση της Ευρώπης είναι ευρωκεντρική. Θα έπρεπε να δούμε τα στοιχεία με μεγαλύτερη προσοχή, αλλά και πιο σφαιρικά, διότι άλλες χώρες δεν τα πάνε αναγκαστικά καλύτερα. Στο φυλάδι που μας δώσατε, εάν κοιτάξει κανείς, τι διαπιστώνει, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε στη Βόρεια Αμερική τέλο πάντων, οι πρόσφυγες είναι 45 εκατομμύρια, 457.000 περίπου. Και αν λάβει κανείς υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών να υποδεχτεί πρόσφυγες, Σκεφτείτε ότι στην Ευρώπη έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες 6 εκατομμύρια στην Αφρική, 3 εκατομμύρια στην Ασία. Βλέπουμε από την πλευρά λοιπόν των δυτικών χωρών ότι η πολιτική ασύλου δεν αποδίδει. Φαίνεται να μην έχει νόημα. Λόγια πολλά ακούγονται για το άσυλο. Στην πράξη όμως δεν φαίνεται να μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το δικαίωμα στο άσυλο. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολλές ε, συνθήκες και πολλές συγκρούσεις μάλλον και συνθήκες πολέμου. Οι πρόσφυγες διώκονται μεν, αλλά στη μισό λεπτό τελείωσα. Στη Λιβύη λόγου χάρη θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό να αποφύγουμε τέτοιε βίε καταστάσει. Ευχαριστούμε κύριε Ζέτα. Ε κυρία Παπαδοπούλου. Κύριε Γκουτέρε, εγώ θα σα καλωσορίσω. Θα πω ότι με έχετε εντυπωσιάσει με τον τρόπο που έχετε θέσει και τα προβλήματα και τι λύσει. Προέρχομαι από την Κύπρο, η οποία είναι επίσης πύλη εισόδου αρκετών αιτητών πολιτικού ασύλου και μεταναστών και λάθρομεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι κύριε Κουτέρες. Εδώ είμαι. Λοιπόν, προέρχομαι από την Κύπρο και η χώρα μου είναι πύλη εισόδου ακριβώς γιατί είναι το νότιο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δέχεται και λαθρομετανάστευση και όταν υπάρχει εμπόλεμο ε, σύραξη στη Μέση Ανατολή ή σε άλλες χώρες, πολλοί πρόσφυγες έρχονται ως αιτητές ε, πολιτικού ασύλου στη χώρα μου. Εμείς όμως βιώνουμε και μια τραγωδία από το 1974 που η γείτονα χώρα η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και δυστυχώς διοχετεύει και ε, αιτητέ πολιτικού ασύλου και λαθρομετανάστε και επίκου παράνομού μέσα από την πράσινη γραμμή στα ελεύθερα εδάφη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η ερώτηση μου είναι συγκεκριμένη. Αναφερθήκατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ολοκληρωμένη στρατηγική και να επιδείξει την κοινοτική αλληλεγγύη. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας όταν μιλάτε για κοινοτική αλληλεγγύη τι ακριβώ πρέπει να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δική μου πατρίδα. Γιατί και εγώ είμαι Ευρωπαία πολίτη και δυστυχώ στερούμε βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μου. Δεν μπορώ να διακινηθώ ελεύθερα. Δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου. Σαν Ευρωπαία πολίτη, τι να περιμένω από την κοινωτική αλληλεγγύη για τη χώρα μου, Ω πρόσφυγα. Um, uh, uh, Ευχαριστούμε. Εδώ, εδώ κύριε εκπρόσωπε. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και σας ευχαριστούμε για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση που έχουμε σήμερα και ευχή όλων μας νομίζω είναι να το συνεχίσουμε και να έχουμε όσο πιο τακτική επαφή μπορούμε. Ε, ξέρω ε, πόσο σημαντική είναι η πατιαρμοστία. Έχω συνομιλήσει πολλές φορές με εκπροσώπους της. Το έζησα όμως και διαζώσεις από κοντά όταν ένα μήνα ε, πριν βρέθηκα στη Συρία ε, όπου είχαμε τη δυνατότητα με, με άλλους δύο συναδέλφους του Κοινοβουλίου, τον κύριο Αγγιλάρ και τον κύριο Ταβάρες, να ε, έχουμε πολλές επαφές εκεί για θέματα προσφύγων. Η Συρία έχει δεχθεί πάρα πολλούς ε, πρόσφυγες εισαγωγικά από το Ιράκ, τους οποίους θεωρεί φιλοξενούμενους, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, νομίζω τα ξέρετε τα θέματα αυτά, είναι πολλά τα προβλήματα και επισκεφτήκαμε μάλιστα και στην Βόρεια Συρία το Al Hol Camp, ένα καταβλισμό για πρόσφυγες, ε, όπου πράγματι η εμπειρία εκεί ήταν πολύ έντονη για όλους μας και γυρνώντας από εκεί και εγώ έτσι ε, ένιωσα αλλαγμένο σαν άνθρωπος και εκεί κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η συνδρομή της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Και πραγματικά το έργο σας είναι κρίσιμο και θέλουμε να έχουμε πολύ τακτική επαφή. Ε, δύο σύντομα σχόλια σε ό,τι αφορά ε, αυτά που είπατε και για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ξέρετε, για όλους εμάς τους Έλληνες δεν είναι καθόλου ευχάριστο να ακούμε ότι στα ζητήματα ασύλου βρισκόμαστε πολύ πίσω. Δυστυχώς όμως και τα περιθώρια τα δικά μας είναι πολύ μικρά. Είναι πάρα πολύ μικρά. Ε, αυτό έχει επιβαρυνθεί και από τη Συμφωνία Δουβλίνο 2 ε, για την οποία θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσά, κατά πόσο πρέπει να την ξαναδούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το ένα λοιπόν είναι για το Δουβλίνο 2, αν νομίζετε ότι πρέπει να ξαναδούμε τη συμφωνία στο εγγύς μέλλον. Το δεύτερο σχόλιο είναι αν πιστεύετε ότι στα πλαίσια της αλληλεγγύης πρέπει να επιδείξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τα θέματα προσφύγων, ε, πρέπει να προωθήσουμε και προγράμματα για reallocation, όχι μόνο resettlement, δηλαδή πρόσφυγες από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, αλλά και εντός της Ένωσης επαναπροώθηση ε, προσφύγων. Και ένα τελευταίο, πώς θα μπορέσουμε... Συγγνώμη, αλλά πρέπει να αφήσουμε στον αρμοστή τον... την ευκαιρία να απαντήσει σε οκτώ σημεία. Σας παρακαλώ, κλείστε. Ε, πώς θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε σε όλους εκείνους που ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον ότι η νόμιμη οδός στην Ευρώπη ε, μέσω ε, των αιτήσεων ασύλου και όλα αυτά που συζητάμε είναι προσφορότερη από την παράνομη μετανάστευση που νομίζω αυτά ε, θα συνδέονται όλο και περισσότερο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you very Ευχαριστούμε κύριε Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει για την κατάσταση διαφορετικών χωρών. Θέλω να δώσω λοιπόν στον ύπατο μα την ευκαιρία να απαντήσει, έστω και σύντομα, σε όλε τι ερωτήσει. Αυτό θα είναι πραγματική δοκιμασία για όλου μα. Έχουμε τρία-τέσσερα λεπτά. Θα προσπαθήσω να είμαι τηλεγραφικό. Και κυρία Ντανόκα, ελπίζω ότι δεν το πρόφερα πολύ λανθασμένα. Το παράδειγμα που δώσατε είναι απόδειξη ότι πρέπει να αναρμονίσουμε τα συστήματά μα. Εάν στη χώρα σα, οι άνθρωποι που έρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση δεν αναγνωρίζονται ω ε, πρόσφυγε και έχουμε πολλού Ρώσου που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, ιδίω από την Τσετσενία, ε, δεν υπάρχει εναρμόνιση και χρειάζεται αυτή. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Οι καταστάσει που αναφέρατε κι εσεί. Οι απάτριδε είναι πρόβλημα. Και είναι και σημαντικό να αναγνωριστούν και τα δικαιώματα των απάτριδων ιδίως στις ε, χώρες της Βαλτικής. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι δεσμευόμαστε και από την Σύμβαση των Απάτρι, για τους απάτριδες. Θα μπορούσε το θέμα να λυθεί άμεσα αν ε, κυρωνόταν η Σύμβαση, αλλά τα δικαιώματα των ε, ανθρώπων αυτών θα πρέπει να γίνονται στο πνεύμα σεβασμού της Σύμβασης αυτής. Η κυρία Αντζελίλη δεν είναι πια εδώ. Απλώ έκανε έκκληση νομίζω για καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό και δεν μπορώ παρά να γρώσω την άποψή τη στην συνάδελφο κυρία Στρέλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Αλλά και σε σχέση με όσα είπατε, ένα κεντρικό ζήτημα στη διεθνή συνεργασία είναι η πρόληψη των βίων μετακινήσεων των πληθυσμών σήμερα. Και να υπάρχει η ε, να δούμε τι γίνεται με τη μαζική προσαρμογή στις ε, μεταβαλλόμενες κλιματικέ αλλαγέ. παγκοσμίω. Ήδη υπάρχουν αλλαγέ, ταχύτατε, ειδικά στην Ανατολική Αφρική, οπότε υπάρχει μαζική κίνηση για προσαρμογή στις κλιματικές ε, αλλαγέ και πιστεύω ότι πραγματικά θα υπάρξουν μετατοπίσεις πληθυσμών λόγω τη απερίμωση ολόκληρων περιοχών που δεν θα είναι πια πρόσφορε για κατοικήσει από ανθρώπου. Στην κυρία Σαρτζεντίνη τώρα για την ε, απέλαση. Νομίζω ότι μίλησε για εσωτερικούς εκτοπισμούς στο Ισραήλ από τη Λορδά της Γάζας. Κοιτάξτε, δεν έχουμε δυνατότητά μας εις παρέμβαση στην περιοχή αυτή. Η να έχει αναλάβει τα, της εκεί περιοχής. Αλλά οι δυσκολίες εκεί είναι διαφορετικών κατηγοριών, θα θυμάστε. Όταν είχαμε τη σύραξη στη Γάζα πριν από λίγο καιρό, η δήλωσή μου ήταν η εξής. Μιλάμε για τη μόνη περίπτωση στον κόσμο όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε πρόσφυγες να γίνουν, δεν μπορούν ούτε να διαφύγουν. Το πρόβλημα λοιπόν που αναφέρατε ξεφεύγει και από την διάσταση των προσφύγων. Βρίσκεται στον πυρήνα του ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχουμε όμως άμεση εντολή εκεί. Και αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα είναι ζωτική σημασίας. Μίλησα για το τόξο κρίσεων. Πιστεύω ότι η επίλυση του ζητήματο τη Παλαιστίνη θα καθορίσει και την επίλυση ενδεχομένω άλλων κρίσεων στον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν, μπορούμε να, δεν είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε προσπάθειε να λυθούν οι υπόλοιπε κρίσει, αλλά αλήθεια αυτή θα διευκολυνθεί η επίλυση των υπολείπων. Η κυρία Φλότρο, να πω ότι το Πακιστάν έχει 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και ίσως να αυτό και λίγο, μου φαίνεται κάπως ηρωνικό μια χώρα που υποδέχεται δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες να έχει τέτοια αιμονή οποιαδήποτε μάλλον χώρα να έχει την αιμονή αυτή να αποστέλει Αφγανούς πίσω στο Πακιστάν. Να, μια χώρα που ήδη έχει το 1,7 εκατομμύρια Αφγανούς στο έδαφος του. Με αυτό το ειρωνικό σχόλιο απλώς να αποπειραθώ να δώσω απάντηση. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να απαντήσω. Για τι ασφαλεί χώρες χώρε τώρα. Υπάρχουν ασφαλώ χώρε οι οποίε δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν ασφαλείς και δεν είναι σίγουρο και το πολιτικό του καθεστώ. Το Μαλί, ε, λόγου χάρη. Υπάρχουμε και, έχουμε και τα προβλήματα του γενετικού ακροτηριασμού. Του γενετήσου μάλλον ακροτηριασμού. Εδώ οι γυναίκες ε, φοβούνται, φοβούνται λόγω της κλειτοριδεκτομής ε, την, πιθανότητα δίωξης στο μαλλί. Πρόκειται λοιπόν ε, για μια πολύ περίπλοκη έννοια. Η έννοια του ασφαλούς τρίτου κράτους είναι πολύ περίπλοκη. Θα προσέξουμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Κυρία Γκυγιόμ, είστε ειδικοί, εκτιμούμε ιδιαίτερως και το έργο που επιτελέσατε ως εισηγήτρια, ιδίως στις τροπολογίες της οδηγίας για τις διαδικασίες για τις δικονομικές διαδικασίες. Οι ερωτήσεις σας νομίζω μόνο με έμεσο τρόπο μπορούν να απαντηθούν. Και είναι και ο μόνος τρόπος να σας απαντήσω με ταχύτητα νομίζω, απαντώντας σας εμέσως. Δώσατε έμφαση στον οικονομικό αντίκτυπο. Είναι κάπως δύσκολο να καταμετρήσει κανείς τον οικονομικό αντίκτυπο στο, εκτός των κατών αυτών. Ε, τώρα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οδηγία για τις υποδοχές σίγουρα θα έχει ένα κόστος, αλλά νομίζω το κόστος αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα συμβαίνουν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιπτώσεις αυτές. Για τον κύριο Κροσέτα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραδεχτούμε ότι οι προσπάθειες ε, για άσυλο τον υπόλοιπο κόσμο, τον αναπτυσσόμενο, είναι εντυπωσιακέ. Ιδίω ακόμη και σε αυτέ τι χώρε που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση του 51 το Πακιστάν. Αυτή τη στιγμή έχει δώσει ταυτότητε, δελτία ταυτότητας, σε 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες που είναι παρόντα στο έδαφος του. Επίσης, πρόσφυγες από τη Συρία και την Ιορδανία επιστρέφουν στο Ιράκ Ε, υπάρχουν λοιπόν ε, δυνατότητες μετακίνησης, κάτι που στο παρελθόν ήταν αδιανόητο. Η Τανζανία έδωσε την επικότητα σε 16.000 ανθρώπους. Κάποιες φορές λοιπόν βλέπουμε οι χώρες των αναπτυσσόμενου κόσμου να έχουν πολύ γενναιόδορη στάση, αν και έχουν περιορισμένους πόρους. Αλλά να μην συνεχίσω με αυτά τα παραδείγματα. Ε, τώρα, κυρία Παπαδοπούλου, αλληλεγγύη μπορεί να υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω είναι πολιτική διάσταση του ζητήματο και αυτό που εσεί αναφέρατε έχει σχέση και με τα όσα ανέφερε ο κ. Παπα-Νικολάου. Δηλαδή, νομίζω ότι οι χώρε στο νότο τη Ευρώπη έχουν αρχίσει να συζητούν ξανά το θέμα τη επανεγκατάσταση, Εδώ Έχουμε δώσει όσα συνεισφορά μπορούσαμε. Εάν υπήρχε εναρμόνιση, θα ήταν καλύτερη κατανομή του βάρου των ευθυνών. Δεν υπάρχει τέλεια λύση. Αλλά νομίζω ότι σοβαρέ προσπάθειε εναρμόνιση μαζί με μια θετικότερη αντιμετώπιση τη κατανομή του βάρου των ευθυνών, ίσω είναι μια λύση. Το Δουβλίνο 2 ζητήσαμε να μην εφαρμοστεί, να μην ισχύει για την Ελλάδα σήμερα, υπό τι παρούσε συνθήκε, και συμφωνούμε και με τις τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή σε σχέση με αυτό το θέμα. Για το τελευταίο ερώτημα, με συγχωρείτε γιατί κάπως έχω χαθεί σε αυτή τη σειρά ερωτημάτων, το τελευταίο σημείο νομίζω ήταν... Δεν μπορώ ούτε να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Τι περίεργο. Υπήρχε επανεγκατάσταση του Δουβλίνο 2 και κάτι ακόμα. What was your last point? Τι είπατε τελευταίο? Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να διαβάσω τι έγραψα. Ε, Πώ ε, ε, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση δίνοντας σε όλους εκείνους που ενδυνάμει θα μπορούσαν να είναι πρόσφυγες το μήνυμα ότι μέσα από την νόμιμη οδό μπορούν να προσεγγίσουν ευκολότερα την Ευρώπη και να μην επιλέγουν τις παράνομες οδούς. Uh, that... Ένα σοβαρό στοιχείο απάντησης είναι το εξής. Μας απασχολεί να διασφαλίσουμε